επόμενη συζήτηση που προβλέπει σύντομη παρουσίαση τη ακόλουθης έκθεσης της κυρίας Λόχ Μπίλερ την καταπολέμηση εμπορία ανθρώπων σε εξωτερικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Συγγήτρια, παρακαλώ για τέσσερα λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη Επίτροπε Μέλστρομ, η μάχη κατά του, της εμπορίας ανθρώπων ε, είναι μια έκθεση πρωτοβουλίας της ε, ε, Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών είναι έργο πολλών επιτροπών έγινε μια πολύ συγκεκριμένη και ειδική έκθεση θέλω να ευχαριστήσω όλες τους συναδέλφους και τους συνεργάτες των εξωτερικών υπηρεσιών το έγκλημα αυτό λέγεται σύγχρονη δουλεία. Υπάρχουν διάφορες ε, μορφές. Ε, υπάρχουν ε, άνθρωποι που θυμίζουν τους αλυσοδεμένους δούλους του παρελθόντος. Ε, υπάρχουν ε, απεισυνασμένοι άνθρωποι που ε, κάνουν σκληρή δουλειά χωρίς αμοιβή ε, και με, κάτω από απάνθρωπες συνθήκες. Ακόμα και σε περίπτωση θανάτου κανείς δεν ενημερώνεται για το δράμα τους. Στην έκθεσή μας ε, αναφέρομαι και μη ορατές μορφές, δηλαδή τα παιδιά στρατιώτες, το εμπόριο οργάνων, ε, καταναγκαστική επαιτία. Ε, όλα αυτά είναι ακραίες μορφές καταναγκασμού ε, που υπάρχουν και δεν μπορούμε να τα καταπολεμήσουμε εύκολα. Ο στόχος εδώ είναι η μέγιστη εκμετάλλευση. Στην έκθεση προτείνω η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη ε, στα διάφορα, στους διάφορους τομείς πολιτικής να ασχοληθούν εντατικά με το θέμα της εμπορίας ανθρώπων ε, φέρνοντας ε, στο προσκήνιο τους θυγωμένους. Θέλουμε ε, οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για αυτή την ε, πέσχεδη κατάσταση να ε, λογοδοτήσουν. Τα θύματα χρειάζονται θεραπεία, βοήθεια, νομική αρρωγή, χρειάζονται αποκατάσταση και αποζημίωση. Η εμπορία των ανθρώπων είναι πολύ επικερδής επιχείρηση και το εμπόρευμα είναι ο άνθρωπος. Οι δράστες αποκομίζουν τεράστια κέρδη. Σύμφωνα με, τον, ε, τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, 150 δις ε, είναι, ε, δολάρια είναι τα κέρδη σε αιτήσια βάση. θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη συνεργασία και με τρίτες χώρες για να στοχεύσουμε τις διαδικασίες ξεπλήματος χρήματος. Οι επιχειρήσεις στο εξωτερικό θα πρέπει να, είναι, ε, να λογοδοτούν για το προσωπικό τους και τις συνθήκες εργασίας του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην εμπορική της πολιτική θα πρέπει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν ούτως ώστε οι συνθήκες ε, να εφαρμόζονται ε, στην πράξη. Οι συνθήκες που προβλέπονται να εφαρμόζονται και στην πράξη. Η Europol και τα κράτη-μέλη θα πρέπει στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος να συνεργάζονται καλύτερα. Και ε, δεν θα πρέπει να ε, περιορίζονται ε, στα σύνορα, οι αστυνομικοί, οι συνοριοφύλακες θα πρέπει να μπορούν να εντοπίζουν καλύτερα τους διακινητές και εμπόρους ανθρώπων είναι πολλά τα μέτρα που μπορεί να βελτιώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αύριο θέλουμε να εγκρίνουμε την έκθεση και χρονικά είναι κατάλληλη στιγμή, ούτω ώστε να επηρεάσουμε την επεξεργασία της, Ευρωπαϊκής, της πολιτικής της Ένωσης για την εμπορία των ανθρώπων. Ε, θέλω τέλος να ευχαριστήσω την ε, κυρία Βασιλιάδου που είναι συντονίστρια ε, στο θέμα αυτό για την εξαιρετική δουλειά που έκανε. Σας ευχαριστούμε κύριε Λόχμπιλερ. Περνάμε τώρα στη διαδικασία Catch the Eye. Δέκα συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο στη διαδικασία Catch the Eye. Ένας ήδη έχει μιλήσει σε τέτοια διαδικασία προηγουμένως. Και γι' αυτό θα ήθελα να περιοριστούμε σε έναν ομιλητή ανά ομάδα. Ο κύριος Μικοάσικ είναι ο πρώτος ομιλητής στη διαδικασία Catch the Eye. Σας ευχαριστώ κύριε Επιτροπέ, κύριε Εισηγήτρια. Ε, η έκθεση ε, της κυρίας Λοχμπιλέρ αφορά την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Ε, μία ιδιαίτερη πτυχή της είναι το εμπόριο ε, ανθρώπινων οργάνων που μάλιστα έχουν εξαχθεί με βίο τρόπο και άνθρωποι που νομίζουν ότι απλώς θα μεταβούν σε άλλη χώρα για ένα καλύτερο μέλλον ε, αντιμετωπίζουν συνθήκες δουλείας. Τα θύματα αυτής της τακτικής πολλές φορές χάνουν τη ζωή τους ε, ενώ τους αφαιρούνται βία όργανα για περαιτέρω μεταμόσχευση στα πλαίσια του εμπορίου οργάνων. Κάτι τέτοιο είναι τελείως ε, αντιφατικό με τη προσέγγιση που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στις εξωτερικές της σχέσεις και στη διεθνή της πολιτική. Σίγουρα θα πρέπει να φροντίσουμε να γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, θα πρέπει η κατάσταση να βελτιωθεί οπωσδήποτε. Ο κύριος Σάνι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση δίνει έμφαση στις διεθνείς πτυχές ε, αυτού του φαινομένου. Δυστυχώς, ε, πολύ συχνά η αυτούργοι της σωματεμπορίας εμπορίας ανθρώπων είναι Ευρωπαίοι πολίτες, ενώ τα θύματά τους είναι γυναίκες και ανήλικοι. οι γυναίκες, τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι είναι πιο ευάλωτες ομάδες, θα πρέπει να έχουν ενισχυμένε προστασίες και φυσικά να μην μείνουν ατιμόρυτοι οι αυτούργοι τέτοιων εγκλημάτων. Θα πρέπει αυτό να αποτελέσει στόχο των εξωτερικών μας σχέσεων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάρεκ Γιούρεκ, χωρίς μικρόφωνο δυστυχώ. Ευχαριστώ. Το εμπόριο ανθρώπων, η σωματεμπορία είναι πολύ σοβαρά θέματα και θα πρέπει να ρωτήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρουμε τι συνέβη με αυτές τις χιλιάδες παιδιά, ασυνόδευτα παιδιά μεταναστών που αγνοούνται. Πού χάθηκαν αυτά τα παιδιά, κάπου στην Ευρώπη χάθηκαν. Αυτή την ε, ερώτηση θέτουμε. Μήπως τα παιδιά αυτά ήταν θύματα ε, εμπορίας ή ε, θύματα για την εμπορία οργάνων. Αυτό το αποτρόπαιο ε, γεγονός μας επισήμανε πριν ο κύριος Μικολάσικ. Ακόμη δεν ξέρουμε πού αγνοούνται αυτά τα παιδιά, ποια ήταν η τύχη τους. Αν πραγματικά ε, λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη αυτό το θέμα, θα πρέπει να συνεχίσουμε να θέτουμε τις ερωτήσεις και να πετούμε απαντήσεις και διαλέφταση. Γιατί θα προκαλέσει κοινωνική διαμαρτυρία αυτό το φαινόμενο. Ε, και πριν από λίγο ακούσαμε από την συνάδελφο πόσο ενδιαφέρεται η κοινή γνώμη για τα θέματα αυτά και πώς τα αντιμετωπίζουμε. Ευχαριστώ. Κύριο Σελίμωβιτς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όλοι συμφωνούμε ότι η εμπορία ανθρώπων όχι μόνο αποτελεί κατάφορη καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελεί και μία μορφή σύγχρονης δουλείας ε, το 2015 και 2016 θα μείνουν στην ιστορία ως οι χρονιές όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι, ευρωπαϊκές, οι εθνικές κυβερνήσεις απέτυχαν να ανταποκριθούν στις ανθρωπιστικές ανάγκες των μεταναστών και προσφύγων που αναζητούσαν ασφάλεια στην Ευρώπη. Αυτά τα δύο χρόνια θα μείνουν στην ιστορία ως οι χρονιές που οι Ευρωπαίοι δέχτηκαν να εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση άνδρες, γυναίκες και παιδιά και να αντιμετωπίζονται ως προϊόντα αντικείμενα συναλλαγή. Χρειαζόμαστε καλύτερο συντονισμό και συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό είναι κρίσιμο και μόνο έτσι θα καταπολεμήσουμε την εμπορία ανθρώπων. Θα πρέπει να δώσουμε μια ρητή και κατηγορηματική απάντηση και πραγματικά να αντιμετωπίσουμε τα θύματα ως ανθρώπους που ε, χαίρουν δικαιωμάτων και να σταματήσουμε αυτά τα εγκληματικά κυκλώματα όσο γίνεται πιο γρήγορα. Σας ευχαριστώ. Η Επίτροπος έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την εισηγήτρια γιατί πραγματικά είναι ένα θέμα που μου είναι ιδιαίτερα προσφυλές. Με απασχολεί ιδιαίτερα και λόγω της προηγούμενης μου ιδιότητας. Φυσικά θα ασχοληθούμε με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων σε εξωτερικές μας σχέσεις και θα προσφροντίσουμε ώστε οι ευρωπαϊκές διατάξεις και οι προδιαγραφές για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων να εφαρμόζονται και θα δώνουμε μάχη παγκοσμίω για υψηλότερες προδιαγραφές κατά της εμπορίας των ανθρώπων, και διμερώς αλλά και σε κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς. Στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, 26 από τις 27 χώρες ήδη έχουν κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή ε, ε, Επιτροπή την πλήρη ενσωμάτωση της οδηγίας κατά της εμπορία ανθρώπων. Μόνο η Γερμανία δεν το έκανε, αλλά μας ενημέρωσε για την πολιτική συμφωνία που έχει ήδη επιτευχθεί και περιμένουμε ε, κοινοποίηση για την ενσωμάτωση τη οδηγία. Στο μεταξύ μένει εκκρεμή η διαδικασία που παραβάσει κατά τη Γερμανία. Στη, στο τέταρτο τρίμηνο του έτους θα υποβάλουμε έκθεση ενσωμάτωση αυτής της οδηγίας και στο πλαίσιο της στρατηγικής του 2006 το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η έκθεση είναι πολύ επίκαιρα. Έχαμε και ένα ορόσημο πρόσφατα το Μάιο με την υιοθέτηση της πρώτης έκθεσης πρόοδου για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Εκεί εντοπίσαμε το μίσο που σημειώσαμε πρόοδο και εντοπίσαμε δυναμίες και κενά στα οποία θα πρέπει να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειές μας. Έχουμε ήδη κάνει πολλά, αλλά πολλά έχουμε ακόμη μπροστά μας. Είναι απαράδεκτο ανθρώπινα πλάσματα να αντιμετωπίζονται ως προϊόντα. Θα πρέπει να σταματήσουμε αυτή, αυτό το φαινόμενο πριν είναι πολύ αργά και να κατατροπώσουμε τα κυκλώματα των λαθρεμπόρων. Θα πρέπει να ενισχύσουμε επίση τη συνεργασία με τι τρίτε χώρε. Η καταπολέμηση εμπορία ανθρώπων αποτελεί τμήμα και τη ε, πολιτική μα μετανάστευση, ε, του σχεδίου δράση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη πολιτική ασφάλεια, καθώ και του ε, πλαισίου δραστηριοτήτων για την ισότητα των δύο φύλων και για τη χειραφέτηση των γυναικών σε εξωτερικέ δράσει μέχρι το 2020. Η διάσκεψη κορυφή Βαλέτα για την μετανάστευση παρουσίασε τη δέσμευση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων για συσπήρωση των προσπαθειών προκειμένου να ε, εξαλειφθεί το φαινόμενο και να παταχθούν ε, αυτές οι πρακτικές και να τιμωρηθούν οι αυτούργοι. Επίσης, ε, θα πρέπει να καταπολεμήσουμε και την λαθροδιακίνηση, αλλά και να αναδείξουμε αυτά τα δύο θέματα, λαθροδιακίνηση και σωματεμπορία, βασικές προτεραιότητες. Ε, σε πολλές ε, συμφωνίες και με τρίτες φορές αναφέρουμε αυτά τα θέματα της καταπολέμησης εμπορίας ανθρώπων, σε διμερείς σχέσεις, σε διαλόγους για ασφάλεια και μετανάστευση και στον διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με 40 χώρες παγκοσμίω ε, αναφέρουμε το θέμα αυτό. Είναι σημαντικό στοιχείο του σχεδίου δράση και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Επίσης στηρίζουμε διεθνείς προσπάθειες στον θέμα αυτό και συμμετέχουμε σε κοινέ δράσεις με πολλά περιφερειακά και διεθνή φόρα όπως ε, ο ΣΑ, ο ΙΕ και ούτω καθεξής. Επίσης θα πρέπει να προωθούμε μια κουλτούρα τιμωρησίας για όσους ε, εκμεταλλεύονται αυτά τα θύματα και να μην αντιμετωπίζουμε τα θύματα ως εγκληματίες. Θέλουμε ισχυρή πολιτική βούληση και δέσμευση και από τους ηγέτες άλλων χωρών. Μόνο έτσι η φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συνδρομή της θα έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο. Και γι' αυτό θα πρέπει να συνεργαστούμε και προσβλέπω στη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρω πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό για σας και ελπίζω να συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Η εμπορία ανθρώπων είναι σχετικά πρόσφατο στοιχείο των εξωτερικών μας δράσεων θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μα, να εδραιώσουμε τα μέχρι τώρα επιτεύγματα και η σχετική έκθεση είναι ένα σωστό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.